Αυτές να είναι οι προτεραιότητες μας και φυσικά να δώσουμε και το βάρος που απαιτείται και στην Ήπεθρο, όχι μόνο στις πόλεις μικρές και μεγάλες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τικάου. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαρθεί αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Μάντερς ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Είναι εδώ η εισηγητής. Very good. Ε, τον λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μάντερς, για τέσσερα λεπτά. Eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο εισηγητής. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν με επιτυχία μαζί μου. Μετά την αυριανή ψηφορία πρόκειται να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας να έχει έτσι το Κοινοβούλιο μία φωνή όταν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι να ωφελούνται οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ. Ελπίζω επομένω ότι όλα αυτά έτσι θα γίνουν. Θέλει τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να δώσει ε, καινούργιες ε, διατυπώσεις στις ονομασίες των ε, υλικών αυτών. Το οποίο ο κύριος Μόντε στην εκθεσή του και μα ανέφερε ποια προβλήματα ανέκυψαν. Τι έγινε με οδηγίες οι οποίες Συνήθω με του κανονισμού εφαρμόζεται κατά 27 διαφορετικού τρόπου. Και εγώ επομένω είμαι όπω ο κ. Μόντι υπέρ του να έχουμε κανονισμού. Και νομίζω επίση ότι οι φάνσιμε είναι, είναι δυνατόν ε, να πετύχουμε καλύτερη ε, πορεία του και μελετήσαμε το θέμα στην Επιτροπή Ιστορική Αγορά και θέλουμε να είναι η διεκπαιρέωση αυτού του θέματο όσο γίνεται πιο αυτόματη. Γιατί αυτό το οποίο εδώ διακυβεύεται για τον Ευρωπαίο πολίτη είναι η, η ονομασία, η ετικετοθεσία όσον αφορά τα είδη ένδυσης. Και εδώ επίσης έχουμε να κάνουμε και με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, άλλο θέμα. Οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε μια αποτίμηση της κατάστασης και να δούμε πώς less is more, πώς δηλαδή με πιο με, λιγότερη νομοθεσία θα πετύχουμε περισσότερα. Με λιγότερα στοιχεία στην ετικέτα θα έχουν περισσότερη ενημέρωση του καταναλωτή. Δεν θέλουμε όμω μια ετικέτα η οποία να αναφέρει τόσα πολλά που να είναι σαν να έχει κανένα κεντήσει ολόκληρη εφημερίδα στο ύφασμα. Θέλουμε επομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε απλές ετικέτες ή στα είδη αυτά, τα κλώστο φαντουργικά. Να ξέρω επομένω όταν πηγαίνω να αγοράσω ένα ρούχο, να ξέρω ε, τι αγοράζω, από πού προέρχεται επίση. Αυτά τα χρειάζονται οι καταναλωτέ. Έτσι θα αποφύγουμε στρεβλέ εμπορικέ πρακτικέ και άδικε. Βέβαια θα πρέπει να καταφέρουμε να ασκήσουμε αποτελεσματικό έλεγχο σχετικά με αυτό. Και να κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα καλύψει την ανάγκη αυτή των καταναλωτών. Εμείς έχουμε διατυπώσει μια σειρά προτάσεων και αφού έχουμε κλωστοφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά 85% στην κατασκευή ενός παιχνιδιού τότε όπως εκεί φροντίζουμε την ασφάλεια των παιδιών, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και όσον αφορά τα στοιχεία που θέλουν να αναφέρονται για κάποιο είδος ένδυση. Αυτό είναι δικαίωμα των πολιτών. Θέλουν να ξέρουν, α πούμε, εάν είναι ζωικό, ζωικής προέλευσης οι ίνες, ε, το υλικό από το οποίο χρησιμοποιήθηκε για, για να φτιαχτεί ένα ρούχο, δέρμα κλπ. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωση κάποιες προτάσεις τις οποίες ενσωματώσαμε εδώ στο κείμενο. Εμείς συμφωνούμε. Ελπίζουμε να μην υπάρχει πρόβλημα με το Συμβούλιο. Θα θέλαμε να υπάρξει αγαστή συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων και να καταλήξουμε σε μια συμβαστική ρύθμιση που να βελτιώσει την κείμενη νομοθεσία και έτσι να μπορούμε να έχουμε τι πληροφορίε που θέλουν οι καταναλωτέ. Ο Σταγιάννη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου για τον θάνατο των δύο Ευρωπαίων στρατιωτών σήμερα το πρωί στο Αφγανιστάν μετά από μια τρομοκρατική επιχείρηση. Κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησε την αναθεώρηση του τομέα της υφαντουργίας στα πλαίσια της ε, βελτιστοποίησης της νομοθετικής δραστηριότητας, της απλούστευσης της νομοθετικής διαδικασίας, όπως επίσης ε, και γενικότερα της διευκόλυνσης των εμπλεκομένων στον τομέα. Θέλουμε έτσι να προωθήσουμε την καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα, να επιτρέψουμε στους κατασκευαστές, στους εμπόρους και στους χρήστες, στους καταναλωτές, να έχουν στη διάθεσή τους νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα με καινοτόμες ίνες. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, όχι μόνο την εφαντουργία, αλλά γενικότερα και την βιομηχανία ένδυσης, φυσικά και, το και τον δημόσιο τομέα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή που υιοθέτησε τη συγκεκριμένη έκθεση την 8η Απριλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντελ και του σκιώδει εισηγητέ για την δουλειά σε βάθος την οποία έχουν κάνει σχετικά με αυτή την πρόταση η οποία οδήγησε σε μια πολύ ζωηρή θα έλεγα συζήτηση γύρω από την ετικετοθεσία των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αρχικό της κείμενο είχε θα έλεγα αποστασιοποιηθεί από τον κανονισμό ο οποίος ήταν υποσυζήτηση τουλάχιστον στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά στο τέλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με τι τροπολογίε τι οποίε είχα παρουσιάσει η Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Συνειδητοποιούμε ότι ορισμένε τροπολογίε, ιδιαίτερα αυτέ, οι οποίε προτείνουν την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού, θα συζητηθούν στο Συμβούλιο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την διαθεσμική, διοργανική μάλλον συζήτηση, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αποδεκτού συμβιβασμού. Μία από αυτέ τι τροπολογίε αφορά το λεγόμενο made in, τη σφραγίδα ή την ένδειξη προέλευσης αν θέλετε. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολλές φορές τον καταναλωτή και είναι ένα θέμα στο οποίο το συγκεκριμένο κοινοβούλιο έχει πάντα δραστηριοποιηθεί με πολύ προσεκτικό τρόπο. Η τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί στην ουσία επαναλαμβάνει την πρόταση την οποία είχαμε κάνει το 2005 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα για τα εισαγόμενα υφαντουργικά προϊόντα. Εγώ θα υποστηρίξω λοιπόν αυτή την τροπολογία όπως είχα τη δυνατότητα να το υπογραμμίσω και στα πλαίσια της συζήτησης με την για την εσωτερική αγορά σχετικά με την τροπολογία η οποία αναφέρεται στην ετικετοθεσία των μη, των μη ε, υφαντουργικών τμήματων, των τμήματων που, προέρχονται από, που έχουν ζωική προέλευση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη προβλέψει συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως επίσης έχει προβλέψει και την εξαίρεση των παραδοσιακών ραπτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ελαφρύνει τις διαδικασίες και ίσως ε, να μπορέσουμε να κάνουμε τις εξαιρέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Θα εξαιρεθούν τις υποχρεωτικής ετικετοθεσίας και θα εξαιρεθούν επίσης και υπερβολικών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Σχετικά με την τροπολογία 63 που θέλει να αφαιρέσει τα παιχνίδια θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ότι το βασικό πρόβλημα για τα παιχνίδια παραμένει το θέμα της ασφάλειας των παιδιών. Η συγκεκριμένη οδηγία έχει επεξεργαστεί σε βάθος το 2009 σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Το θέμα της ασφαλείας λοιπόν έχει αντιμετωπιστεί και από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα παιχνίδια και εμείς ανησυχούμε γιατί το να επιβαρύνουμε τους παραγωγούς έτσι είναι κάτι το υπερβολικό γύρω από το αίτημα της εξέτασης ε, διαφορετικών δυνατοτήτων ετικετοθεσίας για τα υφαντουργικά προϊόντα και προϊόντα ένδυσης. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ευρύτερη συζήτηση από εδώ και πέρα για όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα ακούσω προσεκτικά τις παρατηρήσεις τις οποίες θα κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων πρώτα είναι η κυρία Κόμη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι κομβικός για την ευρωπαϊκή οικονομία η πρόταση την οποία είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια καλή βάση για να βελτιωθεί, αν θέλετε, το διακανονιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα σε επίπεδο διαφάνειας και σε επίπεδο ευελιξίας της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την τεχνολογική πρόοδο την οποία θα πρέπει να επιδεικνύει η φαντουργία. Προσπάθειες τις οποίες κάναμε μέχρι τώρα επέτρεψαν να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυτών υιοθετώντα κανόνες συγκεκριμένους για την ετικετοθεσία που θεωρούμε εμεί απαραίτητη. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή σα στου κανόνε του σχετικού με την ονομασία προέλευση. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάνει δύο προτάσει, δύο συστημάτων διαφορετικών θα έλεγα. Ένα υποχρεωτικό για τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως προεβλέπεται άλλωστε και στον κανονισμό του 2005, φυσικά που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και μια άλλη ετικετοθεσία για τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται στι χώρε μέλη. Έχουμε διητό στόχο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο πρώτος μας και σημαντικότερος στόχος είναι να γνωρίζουμε την πραγματική προέλευση του προϊόντος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να σταθούν ικανοί να κάνουν τις επιλογές τους, ταθμισμένες επιλογές, όταν αποκτούν τέτοιου είδους υφαντουργικά προϊόντα. Μέσω κριτηρίων που προτείνονται θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε οι ετικέτες να περιλαμβάνουν στρεβλές ή παραπλανητικές πληροφορίες εις βάρος του καταναλωτή. Μέσω αυτών των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων θέλουμε να προστατεύσουμε επίσης και τα συμφέροντα των μικρομετέρων επιχειρήσεων που θέλουν να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια εξαρτήθηκε από την επιθυμία που νιώθουμε όλοι να εκφραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι μεγάλες πολιτικές ομάδες. Σε συνεργασία με τον συνηγητή και με τους σκιώδεις εισηγητές ήταν καλή παρότι ξεκινούσαμε από διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς. Συγκλίναμε, καταλήξαμε σε κοινέ θέσεις για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, των πολιτών και του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω αύριο να υπάρξει μια μεγάλη πλειοψηφία και να στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ τον κύριο Μάντες πρώτα πρώτα και τους άλλους που συνεργάστηκαν μαζί του. Ήταν πάρα πολύ θετική η συνεργασία μας για να καταλήξουμε σε αυτό το σχέδιο κειμένο. Έχουμε μόνο τώρα αυτόν τον οργανισμό που θα αφορά τα κλωστοφαντηρικά που είναι μια πρόταση αξιόλογη αλλά και αναγκαία. Νομίζω ότι μας βοηθάει να πετύχουμε εναρμόνιση των διατάξεων σε σχέση με το πώς θα μπορεί να αναγνωρίσει τα νέα προϊόντα στην ε, ενιαία αγορά, τις νέες ίνες. Γι' αυτό και οι σοσιαλιστές είναι υπέρ της ε, πρότασης αυτής. Πάντω το θέμα δεν είναι να βοηθήσουμε μόνο τη βιομηχανία, θα πρέπει να δούμε και το πόσο θα ωφεληθούν οι καταναλωτέ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μα το πώ με αυτή την πρόταση θα εξασφαλίσουμε την ε, ξεκάθαρη ενημέρωση των ε, καταναλωτών σε σχέση με το τι προϊόντα αγοράζουν. Επομένως, θέλουμε να υπάρξει τελικά μια επισήμανση πλήρης όσον αφορά τις πληροφορίες που εκεί θα αναφέρονται. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη σε σχέση με το πώς θα γίνεται γενικά η επισήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, Προσφαντουργικών. Να ξέρει ο καταναλωτής όταν αγοράζει τι αγοράζει, τι περιέχεται εκεί, πού έχουν ε, παραχθεί ε, τα προϊόντα, αν υπάρχουν κάποια αλλεργιογόνα ή στην ίνα και βέβαια και οι συνθήκες παραγωγής είναι σημαντικές. Όλο ένα πιο σημαντικές θα γίνονται στο μέλλον για τους καταναλωτές. Γι' αυτό σα λέω όλα αυτά θα πρέπει να τα μελετήσουμε καλύτερα και να δούμε πώ θα έχουμε τη σωστότερη επισήμανση για τα υπέρ του καταναλωτή. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ τη πρώτη ευθύ κανονισμού. Και προσωπικά πάντως ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνεται με τα διαφορετικά μεγέθη ρούχων ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερε επιδόσει εμπορικέ στην ενιαία αγορά έχοντας τα ίδια μεγέθη για όλες τις χώρες. Και αυτό θα ωφελήσει και καταναλωτές αλλά και την βιομηχανία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, επόμενος ομίλητης τώρα είναι ο κ. Ρινάλντι για φιλελεύθερους δημοκράτες. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή ικανοποίηση για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Συγχαίρω τον κύριο Μάντελς που προσπαθεί να μειώσει την κακοφωνία η οποία ακούγεται ε, στα πλαίσια της συζήτησης αυτής. Σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη προέλευσης και σαν σκιώδης εισηγητές ε, ε, της δικής μου ομάδας, της φιλελεύθερης ομάδας, θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες Κινούμεθα σε ένα διεθνές πλαίσιο παγκοσμιοποιημένο όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στις Ηνωμένε Πολιτείες, στο Μεξικό, στην Κίνα, στην Αυστραλία αλλά και σε άλλες χώρες και αυτό δημιουργεί μια ασυμμετρία και αυτή η ασυμμετρία επιβαρύνει και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκαλούνται δηλαδή κάποιες ίσονες ανομαλίε οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό ισχύει όπως λέγω για τα υφαντουργικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει και μία ποιητική της ένδειξης προέλευσης, κάτι το οποίο επηρεάζει ψυχολογικά τον καταναλωτή και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό. Κινούμεθα σε ένα ομιχλώδες τοπίο ε, μερικές φορές υπάρχει η ένδειξη προέλευσης γιατί βολεύει τον παραγωγό. Κάποιες άλλες φορές δεν υπάρχει η ένδειξη αυτή διότι ο παραγωγός θεωρεί ότι θα λειτουργήσει εις βάρος του εμπορικά. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν, υπάρχουν διαφορές με τις υπόλοιπες χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες και μέσω λοιπόν της προσπάθειας την οποία έκανε ο κύριος Μάντελς και μέσω της προσπάθειας που γίνεται στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προσπαθούμε εμείς να τακτοποιήσουμε κάπως τα πράγματα και να καταστήσουμε το τοπίο πιο διάφανο για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι. Κύριε Ρούλα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον προλαλήσαντα, διότι πιστεύω ότι πρέπει σε αυτό το θέμα να δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή Ίντα, αλλά δεν συμφωνώ με την θέση του μιλητή και σε ορισμένα σημεία δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, διότι πρέπει να τονίσω ότι πρόκειται για το εξή. Όλοι θέλουμε να υπάρχει μια σαφή σήμανση προέλευσης Πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο διότι εδώ και χρόνια ε, έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο αυτή η ονομασία προελεύσεως. Πρόκειται όμως για μια οδηγία και όχι για ένα συμβολικό ψήφισμα. Εγώ είχα στηρίξει μια γραπτή δήλωση η οποία θα απαιτούσε να προχωρήσουμε άμεσα. Αλλά η οδηγία έχει διαφορετικό στόχο. Θέλει να εξασφαλίσει την διαφάνεια για τη χρήση νέων ινών, νέων υλικών και να εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλή τα υλικά αυτά. Όταν θα διευρυνθεί η εφαρμογή αυτής της οδηγίας πολύ φοβάμαι ότι θα έχει την ίδια τύχη που είχε και η προηγούμενη Made In την οποία μπλόκαρε το Συμβούλιο και γι' αυτό πρέπει να δραστηριοποιηθούμε γρήγορα. Συμφωνούμε με όλα τα άλλα θέματα του Made In ανησυχείτε πάντοτε θα είμαστε σύμμαχοί σας αλλά αυτό το ψήφισμα αυτή η ρύθμιση εδώ δεν πρέπει να τη χάνει εκμεταλλεύσεως πρέπει να διορθωθεί ευχαριστώ ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χάρμπορ για δύο λεφτά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απόψε μιλάω για εν ονόματι ε, της κυρίας Μακλόκλιν της ε, ηγητρίας που παρακολουθεί ενεργά αυτό τον φάκελο και ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό που είπε η κυρία Ρούιλε. Συμφωνώ πλήρως μαζί της ε, για το θέμα με το οποίο πρέπει να διεκπαιρεώσουμε το θέμα της ονομασίας προελεύσεως. Γιατί στην πρόταση εδώ έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις σχετικά με την σαφή ουσία της πρότασης όπως θα πρέπει να είναι σαφής η ε, σήμανση και η ετικέτα αλλά αυτό το οποίο δεν ανέφερε ο εισηγητής είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ βασικό θέμα της εσωτερικής αγοράς και της προτασίας του καταναλωτή η οποία αποβλέπει να απλοποιήσει την νομοθεσία να είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε νέα ονόματα και να εισάγουμε πιο γρήγορα νέα υλικά στην αγορά. Ιδίω ε, με την εργασία την οποία κάνουμε σχετικά με την τυποποίηση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα δεδομένα διότι θα περιλάβει όλα αυτά τα θέματα και θα τα προωθήσει στην Επιτροπή Τυποποίησης ε, προς όφελος του καταναλωτή. Βέβαια το ουσιαστικό ερώτημα για τον εισηγητή είναι θέλουμε όλα αυτά τα θετικά στοιχεία να κινδυνεύσουν με το να συνδυάσουμε με την πρόταση αυτή ένα θέμα για την χώρα προελεύσεως το οποίο ήδη ισχύει για πολλά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να μην μειώσουμε τα ωφέλη τα, στα οποία προσβλέπουμε. Βεβαίως πολλά από τα θέματα τα οποία ανέφερε ο εισηγητής πρέπει να προχωρήσουν αλλά νομίζω σε ορισμένα θέματα έχει υπερβεί το ρόλο του σαν εισηγητής της ε, Επιτροπής και προσπάθησε να ε, οικοδομήσει ένα ε, χριστουγεννιάτικο δώρο και να μοιράζει σε όλους δώρα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε αύριο να κάνουμε ορισμένες πολιτικές δηλώσεις, να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές χωρίς όμως να καθυστερήσουμε περαιτέρω. Η κυρία Σπένσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η καταναλωτές πρέπει να μπορούν να επιλέξουν και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μπορούν να έχουν επαρκείς πληροφορίες. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί το πρώτο βασικό δεδομένο για να μπορέσει να προχωρήσει η σήμανση προελεύσεως και να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει διότι έχει δικαίωμα να επιλέξει και πρέπει να έχει σαφείς πληροφορίες. Μετά από αυτό το βήμα βέβαια θα πρέπει να προχωρήσουμε και περαιτέρω διότι θα πρέπει να ε, εξετάσουμε ε, την επεξεργασία, να προειδοποιούμε για τις παρενέργειες, για τις αλλεργίες που μπορούν να προκαλέσουν παραδείγματος χάρη ορισμένα υλικά διότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς για τις υποχρεώσεις και για τη βιομηχανία είναι πολλές φορές δυσνόητες και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να μπορούν να τα καταλάβουν καλύτερα οι καταναλωτές και γι' αυτό χρειάζεται να είναι καλά πληροφορημένοι. Αυτή η έκθεση κύριε Πρόεδρε ονομάζεται και θεωρεί ότι είναι μία μείζον τεχνοκρατική προσπάθεια ε, για να αντιμετωπίσει την κρίση και κάτι που κάνει παραδοσιακά η Κομισιόν όμως και το Κοινοβούλιο προσπαθεί επίσης να χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνοκρατικές εκθέσεις για να μπορέσει να φτάσει σε μια εναρμόνιση και να καταλήξει στο ευρωπαϊκό ή υπερκράτος. Το UKIP θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ ύποπτη εν προκειμένου αυτή η έκθεση. Και εδώ θέλουν να κωδικοποιήσουν και να απλουστεύσουν τρεις χωριστές οδηγίες κατόπιν λένε για κατάργησή τους. Εμείς πάντως το δεύτερο τμήμα το καταδικάζουμε και συγκεκριμένα την τροπολογία 58 εκεί που λέει ότι θα υπάρχει καινούργια επισήμανση που θα πρέπει να εισαχθεί σε επίπεδο ενωσιακό. Και επίση θεωρούμε ότι ε, είναι κακό εκεί που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαία σήμανση των μεγεθών σε υποδήματα και ενδύματα. Εμεί έχουμε μια χαρά σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι τελείω διαφορετικό από το σύστημα στην Πολιτική Ευρώπη οι πολίτες της χώρας μας ξέρουν και καταλαβαίνουν αυτό το σύστημα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δια του εισηγητή του θέλει να χρησιμοποιήσει μια τεχνοκρατική προσπάθεια ούτω ώστε να προωθήσει την αντιδημοκρατική ιδέα του υπερκρατου του Ευρωπαϊκού. Thank you. Ευχαριστώ λέει ο σε χιλιάδες συζητήσεις ε, ε, σχετικά με την παγκοσμιοποίηση φτάνουμε σε ένα σημείο και έχουμε φτάσει στο παρελθόν όπου όλοι αναρωτιούνται τι μέλη γενέστε περαιτέρω και εδώ ανακύπτει η ε, δύναμη και η εξουσία του καταναλωτή ε, και δεν πρέπει κανείς να δυσχεράνει την πορεία αυτή. Ιδίως όσον αφορά τα κλωστοϊφαντουργικά. Αλλά κύριε Επίτροπε, μας λείπει το θάρρος αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για να υπάρξει ένα σήμα. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε για να μπορέσει να υπάρξει διαφάνεια και να ξέρουμε πού και πώς παράγονται αυτά τα προϊόντα, γιατί λυπούμαστε για την έλλειψη θέσεων εργασίας όταν δεν μπορούμε να πούμε στον καταναλωτή τι αγοράζει και πόσο το επιτυχάνει. Ευχαριστώ κυρία Χάντζη, αλλά δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Μάντρες. Ευχαριστώ για την καλή εργασία την οποία κάνατε σχετικά με την ε, ε, οδηγεί αυτή και θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές γιατί εδώ πρόκειται ναι μεν για μία τεχνική έκθεση, επανελήφθη αυτό κατά κόρον, αλλά αυτή η τεχνική έκθεση έχει πολύ ευρείες επιπτώσεις για τους ε, πολίτες διότι πρόκειται για την ε, άδεια κυκλοφορίας ορισμένων ινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όχι όπως όπως πρέπει να τις ελέγξουμε κατά τρόπον ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να είναι ε, σίγουροι ότι υπάρχει προστασία του καταναλωτού την οποία επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι αλλεργιογόνες και πρέπει να υπάρχει και μία σαφής σήμανση κατά τρόπον ώστε ε, οι καταναλωτές και πολίτες να μπορούν να είναι βέβαιοι για το τι αγοράζουν. Στο σημείο αυτό λοιπόν διαφωνώ με τους συναδέλφους οι οποίοι είπαν ότι θα έπρεπε όσον αφορά την ονομασία προέλευσης να την αφήσουμε εκτός. Όχι όμως διότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα κλωστοεφαντουργικά, αυτές οι ίνες, ποιο ε, είναι το παρελθόν τους και το παρελθόν τους είναι εν μέρη και το πώς έχουν κατασκευαστεί με εργασία παιδιών ή με ε, ε, σκλαβιά σε ορισμένες χώρες. Υπάρχουν υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτές τις πληροφορίες για να ξέρουν τι αγοράζουν. Βεβαίως δεν είναι ίσως αυτός ο στόχος αυτής της οδηγίας αλλά εμείς σαν ευρωβουλευτές πρέπει να υπενθυμίσουμε τελικά στο Συμβούλιο και να το πιέσουμε διότι εδώ και ε, δύο πέντε χρόνια από το 2005 πρέπει να καταλάβουμε ότι το κείμενο αυτό πρέπει να προχωρήσει σωστά πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητά του θα πρέπει δηλαδή να εξασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση για να υπάρξει μια σωστή οδηγία ένα σωστό κανονισμός για να μπορεί κανείς να πει ότι ναι αυτό μπορούμε να το δεχτούμε και έτσι να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ενάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένας τομέας βιομηχανικός στην Ευρώπη όπου έχουμε πέσει θύματα αυτών των βίων και βάρβαρων μορφών μετακινήσεων των επιχειρήσεων και κοινωνικού ντάμπινγκ. Η φαντουργία υποφέρει από όλα αυτά. Κάποιες φωλεές θα έλεγα σε πολύ ακριβά προϊόντα υπάρχουν μόνο στην Ευρώπη πλέον και είναι και ιδιαίτερα εύθραυστα όλα αυτά λόγω ακριβώς των παραχαράξεων και κάποιων παράλληλων εμπορικών διαδικασιών. Ό,τι έχει σχέση λοιπόν με την τεχνογνωσία της υφαντουργίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι απαραίτητο. Απαιτείται να υπάρξει και κοινωνική ετικετοθεσία, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέγει επί τη βάση δεοντολογικών θα έλεγα κριτηρίων όπως ε, οι συνθήκες υγιεινής, τα ε, επίπεδα αμοιβή, η κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων κτλ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επίσης την δυνατότητα να καταπολεμήσουμε και την απάτη στα συγκεκριμένα προϊόντα και θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, τις κοινοτικές προτιμήσεις χωρίς να αφήξουμε φυσικά τον τρίτο κόσμο. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόσμπαχ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φαντουργία μέσω ακριβώς της νέας τεχνολογίας και μέσω των καινοτομιών προσπαθεί να επιβιώσει. Ε, βέβαια βλέπουμε ότι πάρα πολλά από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται στην Ευρώπη παράγονται σε χώρες χωρίς κανένα έλεγχο. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στον τομέα της υγείας. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η εναρμόνιση της ετικετοθεσίας ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι και το διαδίκτυο ανήκει νέε ε, ε, ευκαιρίες για τους αγοραστές καταναλωτές. Και γι' αυτό λοιπόν απαιτεί τίτε να υπάρχουν ρυθμίσεις και του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω συγκεκριμένου αριθμού εντοπισμού του προϊόντος, να αναφέρονται ε, ουσίες και χημικές κυρίως ουσίες οι οποίες μπορεί να είναι αλλεργογόνες και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά τα χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί η αγορά. Ευχαριστώ κυρία τώρα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η προστασία του καταναλωτή είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει επομένω να δούμε πώς θα έχουμε κάποιες διατάξεις που κατοχυρώνουν την ενημέρωση του καταναλωτή. Θεωρώ ότι με έναν κανονισμό βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας παρά με τη χρήση των οδηγιών όσον αφορά <coughs> την ενημέρωση για τις σύνες που κυκλοφορούν στην αγορά. Πάντως, συνεχίσουμε και έχουμε κάποια ερωτηματικά που δεν έχουμε απαντήσει, όπως ας πούμε το, τον συνδυασμό ορισμένων συμβόλων ή ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πώς ε, ονομάζεται ο συνδυασμός κάποιων αλλεργιογόνων, προϊόντων τέλο πάντων που αποτελούν αλλεργιογόνα κρίμα, που ακόμα εκκρεμούν αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά δημιουργούν ερωτηματικά όσον αφορά τη χρήση κάποιων προϊόντων. Επίσης, όσον αφορά κάποιε τρίτε χώρε και όσον αφορά από την άλλη μεριά τα προϊόντα των χωρών μελών υπάρχει διαφορά. Και ο καταναλωτή θέλει την ποιότητα, επομένω νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να μπορέσουμε να καλύψουμε με την νομοθετική ρύθμιση και άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι πριν η βιομηχανία μας συρρυκνωθεί, εξαφανιστεί υπό την πίεση των άλλων. Δεν λέω να πάμε σε προστατευτισμό λέω να δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται για συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ενημέρωση είναι μια πραγματικότητα και βελτιώνει μέσα στη, στην παγκοσμιωμένη αγορά την επιλογή του καταναλωτή. Ε, έτσι, επομένως, θα έχουμε πιο συνειδητοποιημένο καταναλωτή. Και είναι δυνατόν να πετύχουμε ποιότητα πληρώνοντας και λιγότερα εργατικά. Γιατί ακόμα, ξέρετε, έχουμε κάποιους ελέγχους που εφαρμόζονται, αλλά δεν γίνονται ισότιμα. Επομένως, πάντως θα πρέπει να επιψηφίσουμε την πρόταση, νομίζω. Ο κύριος Κέλλη τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια προς εισηγητή, προς ε, ε, σκιώδης ε, ε, Προσπαθήσαμε στην Επιτροπή μας να προσεγγίσουμε το θέμα πάντα από την οπτική γωνία του καταναλωτή. Νομίζω ότι εδώ είναι το, θεσμικό όργανο προσέχει περισσότερο τον καταναλωτή της Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που μπήκα στην ιστορική αγορά ε, το, το είδα για τρίτη φορά, για τρίτο νομοθέτημα, το πόσο πιο προοδευτικοί, πόσο πιο ανοιχτοί είμαστε σε σχέση με το, το Συμβούλιο. Ό, όσον αφορά τώρα αυτές τις ονομασίες, όσον αφορά ε, τη, τη, τη, τη σήμανση θα πρέπει να δούμε ότι η προσπάθειά μας ωφελεί και καταναλωτές και βιομηχανία. Είναι προς το συμφέρον επομένως και των δύο αυτή η προσπάθεια. Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι παραγνωρίζει κανείς τα συμφέροντα του καταναλωτή. Τεχνοκρατική προσπάθεια, δεν είναι πολιτική. Προσπαθούμε να κωδικοποιήσουμε τρεις διαφορετικές ε, οδηγίες και επομένως αυτό που θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο είναι να προσπαθεί να καλύψει όσο μεγαλύτερο φάσμα ρυθμίσεων με τέτοιες κωδικοποίησεις. Να έχουμε πληροφορίες τώρα κατανοητές. Να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η σύνθεση του μείγματος, του υφάσματος κάθε φορά να μπορούμε να καλύψουμε τις διαφορετικές ίνες που υπάρχουν στα διαφορετικά προϊόντα, να δούμε πώς θα προλάβουμε κάποια εκδήλωση αλλεργιών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια στις χρησιμοποιημένες μεθόδους. Επίσης, να υπάρχει ακριβή μνήμα τη πρόλευσης. Και έτσι να μπορεί να κάνει την επιλογή τη αγορά του ο καταναλωτής. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούμε να αποφύγουμε στο σημερινό κόσμο προϊόντα που έχουν προέλθει από εργασία ανηλίκων ή καταναγκαστική εργασία. Και νομίζω ότι προσπάθειε νομίζω ότι εμβαθύνεται και στεριώνεται η ιστορική αγορά. Σα ευχαριστώ πολύ πρώτα και τώρα κύριε Μπάστο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μάντελς για μια εξαιρετική προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι τον βοήθησαν στην επεξεργασία της συγκεκριμένης έκθεσης. Πρόκειται για μια προσπάθεια απλώστευσης ε, των ε, κανόνων που είναι ενισχύ και συνδυασμού των τριών οδηγιών που αφορούν την, τον καθορισμό των υφαντουργικών προϊόντων. Η πρόταση αυτή θα επηρεάσει επίσης θετικά νομίζω και τον ιδιωτικό τομέα όπως επίσης και τις δημόσιες αρχές οι οποίες θα μπορέσουν με τη σειρά τους να φροντίσουν καλύτερα την υφαντουργία. Η αναθεώρηση των κανόνων θα βελτιώσει την διαφάνεια των διαδικασιών αδειοδότησης κυκλοφορίας νέων προϊόντων, νέων ινών και νέων ενδυμάτων. Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι παράγοντες δεν έχουν παρά να βρουν πλεονεκτήματα στις νέες αυτές προτάσεις. Νομίζω ότι θα μειωθεί το διοικητικό κόστος και θα υπάρξει δυνατότητα εμπορίας των νέων μορφών ινών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν τις τροποποιήσεις αυτές στην εθνική τους νομοθεσία, κάτι το οποίο θα επιτρέψει φυσικά και περαιτέρω εξοικονόμηση χρημάτων. Και τελικά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία βέβαια είναι ότι ο καταναλωτής θα έχει την βεβαιότητα ότι οι ίνες του προϊόντος θα ε, είναι ε, συμβατές με συγκεκριμένους κανόνες. Επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό, η εισαγωγή νέων ινών είναι απαραίτητη όχι μόνο για την καινοτομία αυτή καθεαυτή, αλλά για τη σωστή προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή. Στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου κόσμου, με τεράστιες αγορές στις οποίες κυκλοφορούν δισεκατομμύρια προϊόντα που ε, παράγονται από εκατομμύρια επιχειρήσεις και βλέποντας την μεγάλη ταχύτητα με την οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κανονισμός αυτός να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν. Μόνο έτσι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και μόνο έτσι θα μπορέσουν να επιδιώξουν νέα τμήματα της αγοράς και θα βελτιώσουν τις συνθήκες απασχόλησης. Κυρία Ράπτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια έκφραση σύμφωνα με την οποία λέμε ότι η ζωή κάποιου ανθρώπου κρέμεται από μια κλωστή. Για φανταστείτε λοιπόν αυτή η κλωστή αν δεν είναι δυνατή, αν δεν είναι από σωστό υλικό, η ζωή θα χαθεί το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό ότι οι κλωστές και τα νήματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι το θέμα μόνο τεχνικό. δεν συζητάμε εδώ μια τεχνική έκθεση. θεωρώ ότι η πολύ καλή έκθεση που έκανε ο κύριος manders και τον ευχαριστώ γι' αυτό έχει μια πολιτική διάσταση μια πολιτική διάσταση που αγγίζει τον έμπορο και τον κατασκευαστή. με τον κανονισμό θα γίνει πιο εύκολη και πιο γρήγορη η δουλειά του μια πολιτική διάσταση που αφορά τον καταναλωτή και κατά συνέπεια την εσωτερική αγορά μια πολιτική διάσταση που αφορά την ηθική πρέπει να ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια του προϊόντος από πού έρχεται. αυτό το made in δεν είναι τεχνικό είναι κυρίως θα έλεγα άκρος πολιτικό όταν ξέρουμε από ποια χώρα προέρχεται ένα προϊόν ξέρουμε πληροφορίες για τον τρόπο που αυτό κατασκευάζεται για τον τρόπο της εργασίας που χρησιμοποιείται εκεί για τα εργατικά δικαιώματα και αν αυτά γίνονται σεβαστά και εμείς εδώ ως πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης δεν είμαστε ε, τεχνοκράτες με κλειστά τα μάτια. είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σκεφτόμαστε νομοθετούμε και ενεργούμε για λογαριασμό των άλλων ανθρώπων. άρα το made in είναι μια τεχνοκρατική ενδεχομένως διαδικασία με μια έντονη πολιτική διάσταση και οφείλουμε πραγματικά κύριε επίτροπε αυτό να το στερεώσουμε σε αυτό νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η δική σας συμβολή. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ήξερα ότι η κυρία Ρούλε είναι πολύ συμπαθητική αλλά μετά από έξι χρόνια επιπλέ, επιτέλους μιλάει στην ψυχή μου διότι αυτή τη στιγμή ε, έχουμε δύο θέματα που είναι στενά συνδεδεμένα και για τους πολίτες ε, και για το Κοινοβούλιο είναι δύσκολο να υποκύψουμε στο Συμβούλιο Πρέπει λοιπόν ε, επιγόντως να βρούμε μία λύση στα προβλήματά μας αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην συνδέσουμε τα δύο διαφορετικά θέματα και πρώτη φορά βλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητάμε για ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ε, λαμβάνουμε αυτό το θέμα και σε ένα άλλο σύνολο που είναι το Made in είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στις επόμενες εβδομάδες ή στην ε, Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Δηλαδή, ε, αν ε, το βαμβάκι έρχεται από το Τουρκμενιστάν, το έχουν επεξεργαστεί στην Νότια Αμερική, από εκεί και πέρα πάει στην Κίνα και γίνεται ύφασμα και ούτω καθεξής, περιπλέκεται το θέμα πάρα πολύ και αν το επιτύχουμε αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό συζητάμε σήμερα αλλά στην εργασία της κυρίας Μουσκαρδίνη και εγώ γι' αυτό θα ήθελα στην δεύτερη ανάγνωση να ε, συνδέσουμε τα δύο θέματα και πάλι και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υποκύψουμε εις ε, το Συμβούλιο και να μπλέξουμε τα δύο πράγματα τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ο κύριος Σούστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή και τους χειώδεις εισηγητές, ευχαριστώ επίσης και τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για τις ε, απαντήσεις τις οποίες ήδη μας έχει δώσει. Εδώ και 18 χρόνια το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης έκανε, ένα, έκανε μια μελέτη και έλεγε ότι η φαντουργία μέχρι το 2000 θα είχε εξαφανιστεί από την Ευρώπη. Ευτυχώς αυτή η προφητεία δεν επαληθεύτηκε για έναν απλό λόγο η έρευνα και η καινοτομία στηρίζουν τις χώρες στις ευρωπαϊκές οι οποίες διατηρούν τέτοιου είδους ε, ε, βιομηχανίες. Δεν ήταν απλά κέντρα ερευνών τα οποία ε, παρήγαγαν προϊόντα, αλλά ήταν εφαρμοσμένη έρευνα μέσα από τις επιχειρήσεις, χάρη ακριβώς και σε μια οδηγία που επιτρέπει στον καταναλωτή να κινηθεί με ευελιξία, ε, να είναι ενήμερος και κυρίως να είναι ενήμερος για την προέλευση του προϊόντος. Νομίζω ότι είναι δυνατόν κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Αντιπρόεδρε Ταγιάννη, να φανταστούμε ένα μέλλον το οποίο να προστατεύει την πρωτοτυπία και τη δημιουργία στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να είναι το θετικό της συγκεκριμένη πρότασης. Η κυρία Γκαρντίνη είναι η επόμενη. Α, εδώ είναι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμεθα τις βασικές γραμμές της πρότασης κανονισμού που βρίσκεται υπό συζήτηση σήμερα, ιδιαίτερα σχετικά με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, την προώθηση της καινοτομίας, και γενικότερα την διευκόλυνση του καταναλωτή και τη σωστή ενημέρωση στον οποίο θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στον καταναλωτή εννοώ. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ε, το λεγόμενο made in. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Ο καταναλωτής θέλει να είναι ενήμερος σήμερα και ακριβώς το να γνωρίσει από πού προέρχεται το προϊόν είναι το πιο ευαίσθητο στοιχείο της ενημέρωσης του καταναλωτή. Αν πάμε σε οποιαδήποτε αγορά, σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης, βλέπουμε ότι οι αγοραστές ενδιαφέρονται στο να αγοράσουν κάτι, γνωρίζοντας όμως τι είναι αυτό, από τι αποτελείται και από πού έρχεται. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πληροφορία αυτή. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται σαν προστιθέμενη αξία. Είναι θα έλεγα σημείο εγγύησης για τον καταναλωτή. Το γνωρίζει κανείς αυτό. Ενώ σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν προβλήματα και το λέμε αυτό χωρίς καμία ε, βούληση ευχαρίστησης. Ε, απλά υπάρχουν κανόνες οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ σωστοί, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι δεν αντιστοιχούν με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, προστασία των παιδιών, συνθήκες εργασίας, σεβασμός των ουσιών που χρησιμοποιούνται. Γενικά πάρα πολλές ειδήσει τον τελευταίο καιρό έφεραν στην επιφάνεια τέτοιες περιπτώσεις, όπως επίσης και περιπτώσεις δυσανεξίας των παιδιών και των γυναικών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προϊόντα. Έχουμε συζητήσει με ιατρούς, με γυναικολόγους, με παιδιάτρους που δείχνουν ότι υπάρχουν αλλεργικές μορφές αντίδρασης σε ουσίες φλαβερές για την υγεία. Δεν μιλάμε για προστατευτισμό εδώ συνάδελφοι. Δεν έχετε άλλο χρόνο λέει ο Πρόεδρος. Έτσι και αλλιώ οι διεθνείς αγορές είναι ανοιχτές και ε, πάρα πολλές χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν τέτοιου είδους ετικέτες. Ο κύριος Σουσβάμπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, σχετικά με τη συζήτηση αυτή την έχω παρακολουθήσει και διαπιστώνω ότι για το ΕΛΚ είναι σημαντικό ο καταναλωτής ο οποίος ενδιαφέρεται για τις πληροφορίες για τα κλωστοεφαντουργικά να τις διαθέτει και ε, γι' αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε ε, τα τεχνικά στοιχεία, να υπάρξει άλλος τρόπος ε, να ε, βρούμε τα στοιχεία. Ναι, ε, το διαδίκτυο είναι χρήσιμο για αυτούς οι οποίοι χρειάζονται πολλές πληροφορίες που δεν υπάρχει λόγος όλες να αναγράφονται ή στην ετικέτα. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές οι οποίοι έθεσαν μία σειρά ερωτήσεων που πρέπει να εξεταστούν αλλά που ε, ε, βέβαια οδηγεί σε μεγάλη αντίσταση για την πρόταση αυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ε, είναι σημαντική αυτή η νομοθεσία ιδίως όσον αφορά τις νέες σύνες οι οποίες όμως δεν θα μπορέσουν να προωθηθούν μέσω αυτού του σχεδίου κανονισμού το οποίο είναι μειονέκτημα για μας και θα έπρεπε τώρα να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας να, το, να επανακτήσουμε την αρχική, το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και να μην τα συνδυάζουμε με το labeling και την ονομασία προέλευσης τα οποία θα εξετάσουμε κάποια άλλη στιγμή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα στη δεύτερη ερώτηση, ε, ανάγνωση οπότε θα εξετάσουμε και τα υπόλοιπα άλλα θέματα τα οποία δεν πρέπει να μας καθυστερήσουν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Σουάμπ. Τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye και βλέπω τον κύριο Σκούρια που θα ήθελε το λόγο. Πήρα το λόγο γιατί θα ήθελα και εγώ να πάρω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Και εμείς βλέπουμε ότι έχουμε εδώ μια πάρα πολύ σημαντική νομοθετική πρόταση. Όχι μόνο για να διευκολύνουμε τις εργασίες των επιχειρήσεών μας, τις δραστηριότητες αυτών, αλλά για να δώσουμε εγγυήσεις στους καταναλωτές έτσι ώστε να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Όποιος επιθυμεί την ποιότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να βρει την ποιότητα αυτή. Πολλές φορές αυτό το οποίο αγοράζουμε πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι αυτό που ονομάζουμε κοινωνικά φόρο, δηλαδή αν έχει ε, γίνει αντικείμενο παραγωγής με σωστές συνθήκες κοινωνικές. Και θα πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα όταν προέρχονται από περιοχές όπου προστατεύεται ο καταναλωτής και ο εργαζόμενος να μην χρησιμοποιούνται παιδική εργασία, να μην χρησιμοποιούνται ε, πρακτικές τρέβλωσης του ανταγωνισμού και θα πρέπει τα μέτρα αυτά να λειτουργήσουν και για άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Θα ήθελα να πω ότι με τέτοιου είδους ρυθμίσεις η Ευρώπη έρχεται κοντά στον καταναλωτή. Και ευχαριστώ τον ε, Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για την προσπάθεια που έκανα. Κυρία Μαγκίνες έχετε το λόγο. Πρόεδρε ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Όλα αυτά τα οποία λέμε τα συζητήσαμε και όσον αφορά τα τρόφιμα, την πρόλευσή τους και την σχετική σήμανση. Ας πούμε μια πίτσα που φτιάχνεται στην Ιρλανδία θα μπορούσε όσον αφορά τα συστατικά να προέρχεται από 60 διαφορετικές χώρες. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να έχει τη σωστή ακριβή σήμανση. Και ένα από τα θέματα το οποίο ότι μας και είναι, είναι να φροντίσουμε οι καταναλωτές να ξέρουν πώς ε, φτιάχνουν τα πράγματα, αν γίνεται σεβαστό περιβάλλον, αν γίνεται σεβαστό το εργατικό δίκαιο. Να, για το CNN έβλεπα ναι, ναι, για κάτι που φτιάχνανε κάτι, κάτι φάσματα εκεί στο, στην Κίνα σε ένα ποτάμι και δίπλα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρήπανση και τελικά αυτά όλα τα εξάγουν πάρα πολύ φθηνά στην Ευρώπη και πάει ο κόσμος και τα αγοράζει. Ε, άρα ο κόσμος θέλει πληροφορίες για να μπορεί ενημερωμένος να αποφασίζει. Πολλοί όμως δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν είναι ενημερωμένοι και αποφασίζουν μόνο βάσει τη τιμή. Άρα θα πρέπει να κοντιάσουν περισσότερο να ευρώ τη βιώσιμη παραγωγή και τη βιώσιμη κατανάλωση. Ε, σε όλο το φάσμα κατανάλωσης για φαγιά όπως και για τα κλωστοφοντουργικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σιλβέστρη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Και εγώ θα ήθελα εδώ να εκφράσω προς την κυρία Ρούλε ε, μια διαφορετική λίγο άποψη. Ε, το λεγόμενο made in λέει ότι είναι υπερβολικό σε, ορισμένους, σε ορισμένες περιπτώσεις να αναφέρεται. Μα τι θα γίνει με όλες αυτές τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στραμμένα, στραμμένα τα βλέμματά τους προς εμάς. Νομίζω ότι ε, δεν θα πρέπει να αποκρύψουμε την χώρα προέλευσης γιατί τότε θα επικρατήσει η Ευρώπη της σιωπή, η Ευρώπη της απόκρυψης, η Ευρώπη που δεν ενημερώνει. Και ε, πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής ε, όχι μόνο το από τι αποτελείται το προϊόν του αλλά και από πού προέρχεται. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει η Ευρώπη της γραφειοκρατίας και του φόβου, η Ευρώπη της σύγχυσης. Θέλουμε λοιπόν να επικρατήσουν οι κανόνες για το Made in και κλείνω πρόεδρε. Αν γράφει το προϊόν Made in Europe, ένα υφαντουργικό προϊόν, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν με τη συγκεκριμένη ετικέτα δεν έχει ε, κατασκευαστεί από προϊόντα τοξικά, δεν έχει κατασκευαστεί, παρασκευαστεί μάλλον από παιδιά, δεν ε, έχουν χρησιμοποιηθεί εργαζόμενοι οι οποίοι σφάζονται από τους εργοδότες τους με ατελείωτα ωράρια εργασίας. Λοιπόν, το Made in Europe είναι εγγύηση για τον καταναλωτή. Είναι εγγύηση και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη ρύθμιση αυτή και να ισχύσει το ταχύτερο δυνατόν. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και ευχαριστούμε και τον Επίτροπο Ταγιάννη για την επιμονή που δείχνει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Νομίζω είναι πάρα πολύ το οποίο συζητούμε τώρα για ένα θέμα το οποίο καίει τον καθένα. Όλους μας. Γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει καταναλωτές και αγοραστές. Και, και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η σήμανση και θυμάμαι πριν από χρόνια ότι πήγα σε ένα μαγαζί και είδα στα Ελλανδικά έλεγε προϊόν Ιρλανδικό. Όμως όταν ε, έβγαλε την ετικέτα είδε ότι από κάτω το αυτοκόλλητο έλεγε Made in China. Επομένως τους γελάνε τους καταναλωτές. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στα του οίκου μας αλλά καθόλου όσον αφορά τα των τρίτων χωρών. Επομένως ε, δεν μπορούμε παρά να χειροκρατήσουμε αυτή την ε, πρόταση. Και βέβαια είναι σωστό να περάσει η πρόταση για ενιαία ονομασία των μεγεθών, παπουτσιών, ενδυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Και καλά μας τα είπε ο κύριος Δούξ, η Βαρόνος τέλος πάντων, για το υπερκράτος, αλλά εν προκειμένου σωστή πρόταση. Ευχαριστώ και τώρα κύριε Φιγκερία, το έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Φιγκερέντο. Έχουμε πάρα πολύ σωστή συζήτηση όσον αφορά την προέλευση αλλά και την σήμανση των κλωστοφαντουργικών. Πολύ σημαντική αυτή η πρόταση υπέρ των καταναλωτών, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τους εργαζομένους, αλλά και την κλώστο στην Ευρώπη. Θέλουμε να καταπονήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά και την εργασία των ενηλίκων. Επίση, θέλουμε να προστατευτούν και τα κοινωνικά δικαιώματα και να πετύχουμε επίση περιβαλλοντική βιομηχανία. Με αυτή τη σήμανση θα μπορούν οι καταναλωτέ να διαλέξουν πάρα πολύ ε, ξεκάθαρα ε, αυτό το οποίο θέλουν και έτσι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μια τέτοια ε, σαφής, σαφούς σήμανση θα φαίνεται το περιεχόμενο του προϊόντος, θα φαίνεται η προέλευση του προϊόντος και θα είμαστε πιο συνειδητοί καταναλωτές και βοηθήσουμε και το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ, λέει ο και όταν γίνει ακούσατε ερωτήσεις, ακούσατε παρατηρήσεις. Μόνο σας δίνω το λόγο για να μας τα πείτε. Συμμερίζομαι και εγώ αυτούς που πιστεύουν ότι αυτή η πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά όχι μόνο. Έχει και σημαντικό πολιτικό βάρος. Έχει πολιτικό βάρος και σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί απλουστεύουμε κανόνες, προσπαθούμε να καταστήσουμε δηλαδή την εργασία του πολίτη, την προσπάθεια μάλλον την οποία κάνει ο πολίτης ε, πιο αποτελεσματική. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Γιατί μέσα από την άποψη που επικρατεί και εδώ στο Κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία της υποχρεωτικής ετικετοθεσίας και σωστής ενημέρωσης, ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τι προϊόν αγοράζει, τι είδους προϊόν αγοράζει, θα μπορεί να προστατεύσει την υγεία του, θα μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά του, τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά φυσικά, και εδώ συμφωνώ με όσα είπε και η κυρία Γκέπχαρτ και όχι μόνο και πολλοί άλλοι ε, ομιλητές και ομιλήτριες. Η προσπάθειά μας είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής υφαντουργίας. Ο τομέας αυτός έχει σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού πολλές φορές. Εμείς θα πρέπει να καταστήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκ νέου ανταγωνιστικές, θα πρέπει να σταματήσουν ε, μορφές dumping στο εσωτερικό της Ένωσης, θα πρέπει να υπερασπιστούμε δηλαδή χιλιάδες θέσεων εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με την προστασία πολλών μορφών και ειδών συμφερόντων συμφέροντα τα οποία νομίζω σέβονται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινωνιών που μας συναποτελούν. Θα ήθελα λοιπόν για το κύριο, αναφέρομαι στον κύριο Ντάρτμουθ, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα υπερκράτος, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Δεν αποτελούμε εμείς τον Λεβιάθαν του Χόμπς. Νομίζω ότι επιδεικνύουμε τις αρχές στις οποίες πιστεύουμε, την αλληλεγγύη, το σεβασμό των ανθρωπίνων αξιών, την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική οικονομία της αγοράς φυσικά και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση εμείς να περιορίσουμε ουδήποτε την ελευθερία απλά να προωθήσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ευχαριστούμε κύριε Πίτρο Πελίο Πρόεδρος και τέλος ο κύριος Μάντρες ο εισηγητής, θα λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι έχουμε για μια τέτοια τεχνολογική έκθεση ένα σωρό παρόντες συναδέλφους Επίσης, βλέπω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση γύρω από την ε, έκθεσή μου. Βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι είχαν επικριτικές παρατηρήσεις για το κείμενο που συνέταξα και είπαν ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία ε, ε, ούτε θα πρέπει να καταχραστούμε και τις οδηγίες που έχουμε ε, ε, περνώντας έναν εικονισμό. Άλλοι είπαν, όπως είπε η κυρία Γκέφχαρτ, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Γι' αυτό πάντω εγώ νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να έρθουν όσο είναι περισσότεροι συνάδελφοι να επιψηφίσουν όσο μπορούν αυτή, αυτή την πρόταση και έτσι να μπορέσουμε στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο να έχουμε μια γερή αφετηρία. Πάντω ευχαριστώ για τι ξεκάθαρε θέσει του τον κύριο Ταγιάννη. Πάντω ε, αύριο νομίζω θα υπάρχει η ατμόσφαιρα που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε μια θέση ισχυρή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ε, νομοπαρασκευή στο μέλλον, να μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτά, το, αυτό το μισό δις καταναλωτών, να μπορούμε να τους δώσουμε τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται. Θα να είναι δυνατόν να κάνει κανένας μια ξεκαθαρή επιλογή. Το θέμα δεν είναι περισσότερε πληροφορίε, είναι το θέμα να υπάρχουν ξεκάθαρε ε, πληροφορίε παντού. Γι' αυτό και χαιρετίζουν πρόταση τη Κομισιόν και επίση θα πρέπει να σα πω, κύριε Πρόεδρε, και να σα υπενθυμίσω ότι εγώ επίτηδε είπα να δούμε τι θα κάνουμε στην πρώτη ανάγνωση. Για να προσέξουμε περισσότερο ως κοινοβούλιο αυτά τα οποία έχει προτείνει η Προσωνή Επιτροπή για την χρηματοοικονομική κρίση. Γιατί η δημοκρατία, ξέρετε, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν κανεί να προκαταλάβει τα αποτελέσματα μια συζήτηση ε, και να τα συμφωνήσει, να τα βρει πριν ολοκληρωθούν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Οπότε δεν πειράζει, α πάμε και σε δεύτερη ανάγνωση να χρειαστεί αλλά ελπίζω πάντως ότι αύριο θα συγκεντρώσω εντυπωσιακή πλειοψηφία για την έκθεσή μου. Εδώ τελειώνει η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος, και θα ψηφίσουμε αύριο για την έκθεση του κυρίου Μάντρας.